Καλημέρα σας συνάδελφοι. Έχουμε πέντε ψηφοφορίες μπροστά μας. Άρα να αρχίσουμε. Πρώτον, έκθεση Βερζιά. Επιστροφή πολιτιστικών εγκαθών που έχουν αποκλειστεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους. Παρένθεση αναδιατύπωση. Ορίστε κυρία Βερζιά, μήπως θέλετε το λόγο ή όχι. Ορίστε. Έχω πει επανειλημμένως ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ νομικού χαρακτήρα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και τους συνεργάτες μας από τις ομάδες που συνεργάστηκαν μαζί μου για την επεξεργασία αυτού του θέματος γιατί Έγινε μεγάλη προσπάθεια αμοιβαίας κατανόησης και σύμφωνα λόγω των συμβιβασμών που πετύχαμε, χάρη στους συμβιβασμούς που πετύχαμε, ελπίζω το τελικό κείμενο να είναι λογικό και συνεπές. Αυτό ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και όλες. Ευχαριστούμε. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ναι, ε? ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση της 16. Έληξε. 7 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται όπως είχα προείπει. Τροπολογία 17 υπέρ κατά πόχες επαλήθευση. Άρχεται, έληξε. 11-11 απορρίπτονται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 1 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 20 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται προφορική 2 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 20 έληξε 15 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται 64 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση. Έληξε 16 με 10 εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται επαλήθευση για την 25 Άρχεται, έληξε. 13 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση 30 επαλήθευση 13 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 10 υπέρ, 15 κατά απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. υπέρ κατά α δεν ήταν σαφές ηλεκτρονική επανάληψη πρώτο τμήμα Δεκατρεις υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ όχι 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ναι, ναι Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. Προφορική 5 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 11 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ υπέρ ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ όχι υπέρ έλειξε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 θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσον ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε άλλη μία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ του να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλειωσε η ψηφοφορία. 23 υπέρ, Άρα δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα λοιπόν πάμε στην έκθεση Camera η έκθεση για την νέα ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ήβα, θέλετε να μιλήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα ε, κυρίως ε, να απευθυνθώ και να ευχαριστήσω τις σκιώδεις εισηγήτρες γιατί ήμασταν μόνο γυναίκες. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή και διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα ότι επί της αρχής συμφωνούμε όλοι και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε την ουδετερότητα των δικτύων στην Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν ότι σήμερα θα καταλήξουμε με ευρεία πλειοψηφία σε μια συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ήτρα ενισχυμένη. Ε, θα είναι σκληρός ο αγώνας για να περάσουμε τη θέση μας. Ελπίζω όμως ότι αν τελικά επιτύχουμε ευρεία πλειοψηφία θα έχουμε όλα τα ατού στα χέρια μας ε, για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με την Ήτρε και να ε, πείσουμε την ε, Ήτρε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα διαδίκτυο δεύτερης κατηγορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Η 82 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ή 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16-84-85 από κοινού υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κλείνει η ψηφοφορία. Πρέπει να αφαιρεθεί μία ψήφος. Ε, να ξαναψηφίσουμε λοιπόν. Ένας από τους φιλελεύθερους δεν πρέπει να ψηφίζει. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. 12 με 13 απορρίπτεται. Η 100 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 105. Ε, υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ η 30 και 107 από κοινού υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. η 32, 110 και 111 από κοινού υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 34. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 113 αποσύρθηκε. Συμβιβαστική 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 124. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 124. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 138 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 38 και οι 139 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, τσίμα τσίμα είναι. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση καλύτερα. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 140. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της 140. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Πρέπει να ελέγξουμε την 140. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται, όπως σας είχα πει. Η συμβαστική 9, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 157. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε την 157. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 160 προφορική δύο υπέρ παρακαλώ. Κατά Δεν ψήφισαν οι φιλελεύθεροι. Ε, προφορική τροπολογία 2 παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 161 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 11 η συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 170 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, γκρίνεται. 172 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήφθηση στην 172. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 173. Υπέρ. Κατά. Επαλήτευση για την 173. Έκλεισε η ψηφοφορία. Γκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 176 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 43 υπέρ, κατά, αποχές πρέπει και πάλι να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 43 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 178 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 182 Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ή 183. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 48. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έκανα ένα λάθος. Πρέπει να επανέλθουμε στην τροπολογία 44. Πρέπει να ψηφίσουμε για αυτήν μαζί με την 190 παρακαλώ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 49. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται μάλλον η 53 υπέρ παρακαλώ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 53 ψηφίζουμε παρακαλώ Έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται Η συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Okay, sorry, compromise 14. in favor? Against, abstain. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 6 και οι 58 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Για την 60 υπέρ, κατά, αποχές. Τώρα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για την 60 παρακαλώ. The vote is closed. Έκλεισε η ψηφοφορία. Into 14, it's rejected. Number 7 and 61, who is in favor. Η 7 και 61 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, γκρίνεται. Τώρα, συμβιβαστική 16. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε την συμβιβαστική 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 17. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 72. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 72. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία εγκρίνεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. η 13 και 18, και 80 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και οι 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια Πέτρα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 Τώρα στην έκτη κυρία Βερχάγκεν. Προετοιμασία για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο. Ζαμπίνε, θε το λόγο? Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της ε, σύνταξη έκθεσης, ε, την πολύ καλή συνεργασία γενικότερα. Σήμερα θα υπάρξουν κάποιες προφορικές τροπολογίες ε, που θα τις λέω όμως όταν θα έρθει η ώρα τους. Ε, θα μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Μπέκερ, ο οποίος επιθυμεί να καταθέσει κάποιες προφορικές τροπολογίες. Έχουμε ένα διαδικαστικό πρόβλημα, διότι δεν είναι δυνατόν να καταθέσει κάποιος προφορική τροπολογία εάν δεν είναι παρόν. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να την κάνω αποδεκτή αυτή την τροπολογία. Yes. Yes. Okay. Okay. Then. Okay. Then we start. Uh, Αρχίζουμε λοιπόν με την ε, τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2, 20 στην 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονική στην 31. Λίγη ψηφοφορία. 10 προς 16 απορρίπτεται. 32. Η Σαμπίνα. Για την 32 θέλω να καταθέσω προφορική τροπολογία. Συγκεκριμένα η πρόταση πρέπει να έχει την εξή διατύπωση. Καλεί την ε, Επιτροπή ε, να ελέγξει ε, κατά πόσον γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας να ελέγχει κανείς το ίδιο το περιεχόμενο να καταρτήσει μέτρα έτσι ώστε στο μέλλον να μην υπάρχει δυνατότητα κατάξυσης. Δηλαδή αυτό που προτείνεται είναι το develop measures, να ληφθούν μέτρα. Πολύ καλά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμ... Με συγχωρείτε. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 στο 53 υπέρ κατά εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 σε δύο μέρη. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στο δεύτερο μέρος της 55. Λίγη ψηφοφορία. 16 προς 9 εγκρίνεται. 56 σε δύο, σε χωριστή. Στο πρώτο μέρος, υπέρ, η Ζαμπίνα αυτό ο κύριος Μπεκέ απέστειλε το Satchel TV Alliance που σημαίνει ότι επ' αυτού δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Άρα δηλαδή μόνο μία ψηφορία για το 56. Εντάξει λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58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 Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77. Ε, με συγχωρείτε, 78. Υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. 79. Υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. 80. Υπέρ, κατά, αποχές. Με συγχωρείτε, κατά, ποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην 80. Λίγη ψηφοφορία. 17 προς 12 εγκρίνεται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κυρία Χέρσου. Θα ήθελα να προσθέσω και μια προφορική τροπολογία. Να προσθέσω στην πρόταση όπου υπάρχει πρόσβαση και μπορεί κανείς στον σημερινό κόσμο να βρει την χρήση των οπτικοακουστικών μέσων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 15 προς 14, εγκρίνεται. Στην 8 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Πρώτη υπόδειξη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 9 ε, ναι, προς 20, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. 6. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 7 ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερον μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, συνάδελφοι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 17 προς 11. Υπόδειξη 8. Το πρώτο. Μέρος υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ ηλεκτρονική. ηλεκτρονική. Λίγη ψηφοφορία. 26 υπέρ και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια Ζαμπίνε. Λοιπόν, περνούμε τώρα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν κόσμο στον οποίο επικρατούν πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές. Θέλετε το λόγο κύριε Παπα-Νικολάου? Όχι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία. 10 προς 17. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται το τέταρτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά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 Λίγη ψηφοφορία. 15 προς 10 εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση στην 43, παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία. 15 προς 14. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση.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 Θέλετε, Λόκεγκαρντ, το λόγο. Ας αρχίσουμε. Πρώτη τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερον, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 σε τρία μέρη. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δέκα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έντεκα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ε, ψηφοφορία, συγγνώμη. Ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. 27 με μία εποχή Κύριε Λόκεγκαρτ, συγχαρητήρια.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο όπου υπάρχει τόσο ψηλή ανεργία και ιδιαίτερα των νέων. Από την άλλη βλέπουμε μια κατάσταση όπου υπάρχουν πολλές κενές θέσεις απασχόλησης γιατί δεν έχουν οι ενδιαφερόμενοι την απαραίτητη κατάρτιση. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι διδάσκουμε στους νέους στα σχολεία μας. Πόσο έτοιμοι είναι αυτοί οι νέοι να μπουν στην αγορά εργασίας όταν βγουν από το σχολείο. Διότι από τη μία υπάρχουν οι ανάγκες των εταιριών και επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας και απ' την άλλη η διαφορά με τις δεξιότητες που μαθαίνουν οι νέοι στα σχολεία. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για, για την πολύ ψηλή ανεργία ιδιαίτερα των νέων. Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και ανοιχτή πόρη εκπαίδευσης μπορεί να είναι ένα μέρος της λύσης στο πρόβλημα, διότι έτσι δημιουργούνται νέες δεξιότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας και απ' την άλλη διευρύνονται πολύ οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για τεκμηρίωση και διδασκαλία και μάθηση και αποτελούν διαδραστικές και εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές πραγματικότητες. Βέβαια δεν είναι εύκολα όλα αυτά γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για την θέληση των νέων να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους αλλά για πολύ ουσιώδεις επενδύσεις που χρειάζονται για να μετεκπαιδευτούν οι δάσκαλοι οι ίδιοι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους, να ε, ασχολούνται με νέα θέματα εκπαίδευσης που να τα διδάσκουν με τελείως διαφορετικό τρόπο διότι εδώ μιλάμε για διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και πόρους που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προφανής η χρησιμότητά τους και το περιεχόμενο πρέπει να είναι παρόμοιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα ποιος θα σχεδιάσει αυτούς τους εκπαιδευτικούς πόρους, ποιος θα αποφασίσει αν και πώς ε, και κατά πόσον ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν σε όλες τις χώρες μέλη. Βέβαια, ένα εκπαιδευτικό, μια εκπαιδευτική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει ένα νέο να μπει στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και πρόβλημα αν ανταποκρίνεται μόνο στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Είναι λοιπόν μεγάλη η πρόκληση, αλλά αυτό είναι το μέλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ μελλοντική παιδεία χωρίς τη χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, το ίντερνετ κλπ. Είναι γεγονός ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχουν όμως ορισμένα καλά παραδείγματα όπως στη Σλοβενία όπου σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Μίλησα με τον Υπουργό Παιδείας της Σλοβενίας και μου είπε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα πειραματικό επιλοτικό πρόγραμμα <clears throat> με βάση τη Σλοβενία που να χρησιμεύσει τελικά για τη διάδοση βελτίστων πρακτικών πανευρωπαϊκών. Βέβαια αυτό το νέο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει και όσους θέλουν να βελτιώσουν απλώς τις δεξιότητές τους, οι λιγότερο νέοι δηλαδή, που δεν είναι πλέον φοιτητές να χρησιμοποιηθεί δηλαδή και για τη διαβίου μάθηση που θα βελτίωνε Την οικονομική τους κατάσταση. Αυτές οι νέες μέθοδοι λοιπόν με μεγαλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορία είναι πιο, πιο εύκολη. Φυσικά μπορεί κανείς να την κάνει και από το σπίτι του, δεν χρειάζεται να οδηγήσει 100 χιλιόμετρα για να πάει σε κάποιο σχολείο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όσοι είναι 30, 32, 34 ή 50 ετών δεν γνωρίζουν πολύ καλά ίσως τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. <clears throat> Να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για καμπή στην ιστορία της παιδείας. Για ένα χρονικό σημείο όπου σημειώνεται η μετάβαση, δηλαδή δεν εγκαταλείπουμε τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά υπάρχει μια μετάβαση προς ένα μείγμα, ε, μια μίξη και των παραδοσιακών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών. Όσοι σπούδασαν αποκλειστικά με το παλαιό σύστημα, ίσως όμως να έχουν πρόβλημα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Και τέλος, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να στηρίξουν και απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Την Ελλάδα την αναφέρω γιατί έχει πολλά νησιά νησιά όπου είναι λίγα τα παιδιά και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οργανωθούν εκεί σχολεία ή να μεταφερθούν τα παιδιά από το ένα νησί στο άλλο. Ο ευκολότερος τρόπος για να παρακαμφθεί αυτή η απομόνωση είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας με πλασματικές τάξεις, με διδασκαλία online ώστε και οι μαθητές από αυτές τις απομακρυσμένες κοινότητες να υποφελούνται, όποια και να είναι η απόσταση μεταξύ δασκάλου και μαθητού. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να οργανωθεί μόνο, πανενωσια, μόνο από την Ένωση αυτό, αλλά και τοπικά και περιφερειακά. Μιλάμε για υπερνίκηση της κρίσης για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Αυτό όμως σημαίνει αναγκαστικά ότι θα έχουμε μια πολύ καλά ένα πολύ καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και θα μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται στις καινούργιες συνθήκες της σύγχρονης οικονομίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί ζητούμε μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά η επιτυχία θα μετρηθεί από το κατά πόσον μπορεί κανείς πρώτα να δημιουργήσει μια καλά, ένα καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό όσο το δυνατόν κοντύτερα στην ε, κατοικία του ο καθένας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει η οικονομική υποστήριξη της νέας αυτής τεχνολογίας για την εκπαίδευση να προέρχεται και από τις επιχειρήσεις και από την Ένωση και από τις τοπικές αρχές. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε τα πανεπιστήμια ώστε να δημιουργήσουν κοινά προγράμματα, κοινά προγράμματα γιατί θα ήταν πάρα πολύ θετικό να μοιραστούν τα πανεπιστήμια αυτές τις ιδέες και μεθόδους. Αργότερα, αν χρειαστεί, θα επανέλθω αυτά. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι χτες ε, συζητήσαμε διεξοδικά για το θέμα αυτό με τους εμπειρογνώμονες Άρα δηλαδή ε, σήμερα δεν θα θελήσουν πια οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Ε, άρα δηλαδή αυτά που είπαμε χτες τα στηρίζουμε και στηρίζουμε επίσης ε, το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς οι οποίοι για καθαρά γεωγραφικούς λόγους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε σχολές περαιτέρω κατάρτισης, σε καλύτερη εκπαίδευση, ότι όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αναφερθήκατε στα νησιά, αλλά αν δείτε λιγάκι την μορφολογία του εδάφους ε, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, όπου δεν υπάρχουν ε, οι απαραίτητες αστικές κοινωνίες, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα νέα μέσα. Εχθές ε, δεν συζητήσαμε γι' αυτό, συζητήσαμε περισσότερο για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, νέες τεχνικές χωρίς να αντικαταστήσουμε τις παλιές. Και το πρόβλημα είναι, το είπαμε αυτό και χθε, ότι δεν είμαστε σε θέση να αναγκάσουμε κάποιον να χρησιμοποιεί τις νέες δυνατότητες. Αυτό είναι καθαρά εθνικό θέμα και νομίζω ότι εμείς με τις ε, προτάσεις μας το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, προσφέρουμε κίνητρα. Εγώ λοιπόν εύχομαι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων να προσφερθούν οικονομικές δυνατότητες έτσι ώστε κυρίως σε αγροτικές περιοχές, σε υποβαθμισμένες περιοχές ε, να ε, μπορούμε να προσφέρουμε κάποια βοήθεια. Ε, συζητήσαμε διεξοδικά για χτες γι' αυτό. αν κάποιος θέλει να λάβει παρόλο το λόγο, παρακαλώ. Αλλά όπως σας είπα, ε, Εχθές συζητήσαμε διαμακρών για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σήμερα. Μήπως θέλετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείτε κάτι, παρακαλώ. Εξ ονόματος της Κομισιόν θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που αποφάσισε να συζητήσει και αυτό το θέμα η ανακοίνωση που κάναμε πρόσφατα δείχνει ότι και η Κομισιόν έχει καταλάβει τη σημασία που έχει χρήση αυτών των τεχνολογιών για την παιδεία σε όλες τις, τις πτυχές. Την πρόσβαση, την ψηφιακή καθυστέρηση, αλλά Επίσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παιδείας που να μπορεί να γίνει με τρόπο πιο προσωπικό, πιο προσαρμοσμένο ως στις ανάγκες του καθένα ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά του. Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο που συζητά αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε. Ο Ήβαν. Εχθές έπρεπε να πάω στη συνεδρίαση των σπιωτών αλλά δεν μπόρεσα δυστυχώς γιατί έφτασα μόλις σήμερα το πρωί μόνο και μόνο για να σας μιλήσω εδώ. Θα ήθελα να κάνω ένα μόνο πρόσθετο σχόλιο. Ό,τι σχετίζεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όπως στη δημιουργία προγραμμάτων μάστερ, μαθημάτων μάστερ στα πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να είναι όλα δωρεάν εφόσον χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά χρήματα. Οι ιδιωτικοί πόροι που χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια είναι άλλο θέμα, αλλά οτιδήποτε χρηματοδοτούμε εμείς πρέπει να είναι δωρεάν για τους πολίτες. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος, θα το λάβουμε υπόψη μας ε, και θα το δείτε και μετά στις εκθέσεις που θα δημοσιευτούν. Να σας πω ότι την 3η 6 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την έγκριση των ε, τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου Ήβαν. Έτσι λοιπόν ε, με αυτό το θέμα εξαντλήσαμε σήμερα την ημερήσια διάταξη και περνάμε τώρα στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών και όσοι δεν έχουν σχέση με τους συντονιστές αν θέλουν να πιούν καφέ ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. μην ξεχάσετε όμως ε, το απόγευμα να έρθετε όλοι, μην έχουμε εδώ άδεια αίθουσα. Τρεις υπουργούς θα έχουμε, τρεις υπουργούς από την Ελλάδα. Και δεν μ' αρέσει να έχω άδειε καρέκλες μπροστά μου. Ευχαριστώ.